Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, περνάμε τώρα ε, στη μυστική ψηφοφορία για ορισμό μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για τον ε, ορισμό του κυρίου Νέβεν Μίμητσα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ κατά αυτού του ορισμού. Δεν θα λάβει κανείς τώρα το λόγο. Ψηφίζουμε με μυστική ψηφοφορία Κατόπιν τούτου θα ανάψει μόνο το μπλε φως, για να μην ρωτάτε το λέω αυτό, αν θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε όχι ή αποχή, αλλά σας επισημαίνω ότι θα ανάψει μόνο το μπλε φως. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Ρωτάω λοιπόν, εψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. ...565 υπέρ, 64 κατά και 64 αποχές. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μίμητσα ορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής. Το λόγο έχει ο κύριος Ρεν εκ μέρους της Επιτροπής. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Ρεν. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συμβάσεω Προσχωρήσεω τη Κροατία Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο διαβουλεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ψηφοφορία που μόλις έγινε εξέφρασε την θετική άποψη του Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόθεση του Συμβουλίου να ε, ορίσει σε αυτήν τη θέση την κυρία Μιμιτζά. Εμεί εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση και τώρα θα πρέπει το Συμβούλιο να συμφωνήσει με τον πρόεδρο και συντροπή ώστε να γίνουν τα τελευταία διαβήματα για αυτόν τον ορισμό. Εμεί ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο που ολοκλήρωσε την ε, ε, διαδικασία της διαβούλευσης που έγινε αποτελεσματικά και έτσι μπορέσαμε και εμείς να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ε, της πρόσχολης της Κροατίας αρχές Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ ε, τον Επίτροπο μάλλον και ψηφίζουμε τώρα για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων Συνόδου του Κοινοβουλίου 2014. Το λόγο έχει ζητήσει η κυρία Λούλινγκ. Euh, euh, euh, Εν συντομία, να σας ε, εξηγήσω γιατί έχω υποβάλει μια τροπολογία μαζί με άλλους συναδέλφου και να σας ε, ενημερώσω ε, προκειμένου να μην ψηφίσουμε ένα παράνομο χρονοδιάγραμμα. Η τροποπιλογία δεν είναι πολιτική, είναι νομικής φύσεως. Δεν ψηφίζουμε υπέρ κατά της σκοπιμότητας να έχουμε στι της Ε, Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι αποφάσει του δικαστηρίου, για παράδειγμα του Δεκεμβρίου 2012. Αν δείτε το χρονοδιάγραμμα, το ημερολόγιο που έχετε μπροστά σα, θα δείτε ότι περιλαμβάνει 11 ολομέλειες στο Στρασβούργο. Ε, η συνθήκη καθορίζει 12, αλλά η πρακτική είναι σε χρονιά εκλογών να έχουμε 11 Ολομέλειες ε, στο Στρασβούργο. Αυτό το έχει δεχτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με ε, δεχόμενη την, δεχόμενο την εξαίρεση αυτή για τις εκλογικές χρονιές. Όμως το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Το Δεκέμβριο 2012 με απόφαση του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο σημείο 57 αναφέρει ότι οι πρόσθετες ολομέλειες σύνοδοι μπορούν να οργανωθούν μόνο αν ε, προβλέπονται 12 ολομέλειε στο Στρασβούργο. Αυτό είναι λογικό. Δεν είναι δυνατόν από τη μια μεριά να λέμε ότι 12 είναι πολλές στο Στρασβούργο για την εκλογική χρονιά και από την άλλη μεριά να αποφασίζουμε πρόσθετες ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Συνεπώς έχουμε την επιλογή είτε να οργανώσουμε 11 ολομέλειες στο Στρασβούργο και καμία στις Βρυξέλλες ή να οργανώσουμε 12 ολομέλειες στο Στρασβούργο οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προβλέψουμε και πρόσθετες, τρεις πρόσθετες ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Συνεπώς, ή 11 στο Στρασβούργο και καμία στις Βρυξέλλες ή 12 στο Στρασβούργο και τρεις πρόσθετες ολομέλειες. Αυτό για να καταλάβουν οι συνάδελφοι και ε, να μην υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα προτείναμε λοιπόν εμείς την πρώτη λύση. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε και τη δεύτερη. Αλλά προτείναμε την πρώτη. Αν δεν συμφωνήσετε, δεν συμφωνήσει το σώμα με την πρότασή μας, το ημερολόγιο, το χρονοδιάγραμμα του 2014 ε, μπορεί να γίνει αντικείμενο προσφυγής στο, Ευρωπαϊκό, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφύγουμε αυτή την ε, οδυνηρή ε, περίπτωση θέλησα να σας εξηγήσω την τροπολογία και να σας ζητώ να την υπερψηφίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λούλινγκ, κατόπιν του, του κυρίες και κύριοι. Ε, παρακαλώ την προσοχή σας για λίγο. Κυρία Λούλινγκ, άκουσα προσεκτικά αυτά που μας ε, είπατε. Ε, προφανώς συζητήσαμε διαμακρών όσον αφορά την τροπολογία αυτή, κατά πόσο είναι αποδεκτή ή όχι. Και αποφασίσαμε ότι είναι αποδεκτή. Οι 12 ολομέλειες στις οποίες αναφερθήκατε το 2012 ε, δεν ήταν αντικείμενο αποφάσεων για εκλογικά έτη. Το ε, δικαστήριο όσον αφορά τα εκλογικά έτη αποφάνθηκε και το δικαστήριο αναφέρει ότι είναι επιτρεπτές 11 συνεδριάσεις διότι οι 5 ημέρες οι οποίες κρίνονται ως ημέρες εκλογών. Αυτές οι ημέρες προσμετρώνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα σε τέτοιου είδου έτη υπάρχουν μόνο 11 ολομέλειες. Άρα δηλαδή κατά αυτά τα εκλογικά έτη επιτρέπεται να ε, υπάρχουν περισσότερες ολομέλειες Βρυξέλλε. Και γι' αυτό λοιπόν ψηφίζουμε τώρα. Ε, υπέρ του, της πρώτης τροπολογίας παρακαλώ ψηφίζουμε κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα δηλαδή εγκρίνεται αυτό ε, και κατόπιν τούτου έκλεισε το θέμα του ε, ημερολογίου, αλλά τώρα θα διακόψουμε για να έχουμε ε, την πανηγυρική εκδήλωση με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας, τον κύριο Καβάκο Σίλβα και είσαστε όλοι θερμά προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση αυτή.